Καλημέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους της σημερινής συνεδρίας τη Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των αντιπλωματικών αποστολών, ιδίως την αυτοεξοχότητα κύριο Αλφάρο, πρέσβη της Κωνσταντίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αυτοεξοχότητα τον κύριο Μανδρίτ, πρέσβη της Ονδούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καλωσορίσω επίσης τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν, τον κύριο Νταλιρίτσια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την κυρία Λολίτα Μπουτκεβίτσιενε, προϊσταμένη της Μονάδας για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, Επίσης, να καλωσορίσω τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, την κυρία Γιάκομσεν, μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, και να σας πω ότι η διερμηνία παρέχεται στα αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά, πορτογαλικά και πολωνικά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης Δεκεμβρίου του 2016 περιλαμβάνονται στο φάκελο και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης ε, θα εγκριθούν χωρίς αλλαγή. Και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σα ενημερώσω σχετικά με την πορεία των εργασιών για τη σύσταση τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική. Η γραμματεία τη μονάδα τη Λατινική Αμερική ήρθε σε επαφή ξανά με του ομολόγου τη στην Εθνική Συνέλευση τη Κώστα Ρίκα πριν από τα Χριστούγεννα και ρώτησε σχετικά με την διαδικασία επιβεβαίωση των αλλαγών στον κανονισμό τη διαδικασία που προτείνει το Παρλασέν. Οι προτινόμενες αλλαγές αφορούν στην κατανομή των εδρών του στοιχείου της Κεντρικής Αμερικής στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των κανονισμών, και η Εθνοσυνέλευση μας διαβεβαίωσε, διαβεβαίωσε τη γραμματεία μας ότι θα λάβει απόφαση αμέσως μετά τις διακοπές του τέλους του προηγούμενου έτους. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σε επαναλάβω την αποφασιστικότητά μου να καθοριστεί η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτου. Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω ότι το Δεκέμβρη ο τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σούλτ έλαβε ένα γράμμα από την πόλη Σουανή όπου τον ενημέρωναν σχετικά με την υιοθέτηση τη απόφαση καλέσματο για την άμεση απελευθέρωση τη κυρίας βάσκε πολίτη του Ελ Σαλβαδόρ. Η κυρία Βάσκε είναι μια ακόμη γυναίκα που τιμωρείται στη βάση των αυστηρών κανόνων κατά των αμβλώσεων που ισχύουν στο Ελ Σαλβαδόρ. Το 2008 η κυρία Βάσκες καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για βεβαρημένη ανθρωποκτονία αφού υπέστη θνησιγωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Στο Ελ οι γυναίκες που αποβάλλουν ή υπόκεινται θνησιγένεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνήθως γίνονται οι υποπτές ότι έκαναν έκτρωση. Η έκτρωση κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες είναι ένα έγκλημα, ακόμα και σε περιπτώσει βιασμού, αιμομηξίας ή όπου η ζωή μια γυναίκα είναι σε κίνδυνο. Το γεγονό αυτό καθιστά τι γυναίκε φοβισμένε στο να ζητήσουν βοήθεια για προβλήματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, οδηγώντα αναπόφευκτα σε περισσότερου θανάτου που είναι αποτρέψιμοι. Η διεθνή Αμνηστία έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για την απελευθέρωση της κυρίας Βάσκες και μπορείτε να βρείτε την επιστολή, της, την επιστολή αυτή στα αρχεία σα. Περιμένουμε την απάντηση που θα δώσει ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο θέμα του, του σχεδίου χρονιαδιαγράμματος και δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάμεινο του 2017. Στο φάκελό σας, σας έχει που σας έχει διανεμηθεί θα βρείτε το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της αντιπροσωπείας για το δεύτερο εξάμεινο του 2017 που όπως θυμάστε είχαμε συζητήσει πέρσι την πιθανότητα επίσκεψης της αντιπροσωπείας στην Κούβα μέσα στο 2017. Μετά την υπογραφή τη Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κούβα στι 12 Δεκεμβρίου του 2016, μία επίσκεψη πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Κούβα. Είμαι σε συνεχή επαφή με την, με την κουβανική πρεσβεία για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την οριστική απάντηση από την κουβανική πλευρά σχετικά με την έγκριση αυτής της επίσκεψης. Το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην ανταλλαγή απόψεων για τους στόχους της προσωρινής Προεδρίας της Κώστα Ρίκα του Συστήματος Ολοκλήρωσης Κεντρικής Αμερικής για το πρώτο εξάμεινο του 2017. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, στις 20 Δεκεμβρίου του 2016 η Κώστα Ρίκα ανέλαβε προσωρινά την Προεδρία του Συστήματος Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Κώστα θα πρέπει να κατευθύνει την κεντροαμερικανική κοινότητα σε εποχές που προμηνύονται ταραχώδεις και σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Η ΣΥΚΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες ή άμεσες προκλήσεις που θα τεθούν από τη διοίκηση Τραμπ στις ΗΠΑ, διότι όπως γνωρίζετε οι επιπτώσει των νέων πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό θα γίνουν αισθητέ και στις γειτονικέ χώρες. Παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις που πρόκειται να συμβούν, η Κώστα θα καθοδηγήσει επίσης τη ΣΥΚΑ σχετικά με το ζήτημα του μετασχηματισμού του θεσμικού συστήματός της. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι η Κώστα Ρίκα είχε αποσυρθεί από τον πολιτικό πυλώνα του ΣΥΚΑ το Δεκέμβριο του 2015 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση από άλλες χώρες να συνεργαστούν για την εξέβρεση λύσης στην κρίση της μετανάστευσης. Την 1η Ιουλίου του 2016 η κυβέρνηση της Κωνσταντίνα ανακοίνωσε την επιστροφή της στη ΣΥΚΑ έπειτα από τη δέσμευση των χωρών μελών ότι θα εργαστούν για ένα σοβαρό, αμφιχτικό και διαφανές σύστημα ολοκλήρωσης. Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση έχει εργαστεί σε μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του ΣΥΚΑ, η οποία θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην περιοχή με ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη τι έκτακτε προκλήσει που προκύπτουν το διάστημα αυτό, χαιρετίζω θερμά την ανακοίνωση τη Κώστα Ρίκα και του Παναμά, που θα αναλάβει την προσωρινή προεδρία τη ΣΥΚΑ για το δεύτερο εξάμεινο του έτου, για το στενό συντονισμό των εργατιών του, και θα δώσω αμέσω το λόγο στην αυτοεξοχότητα τον κύριο Αλβάρο, πρέσβη της Ρίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μα ενημερώσει. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Και σε γενικές γραμμές να σας ευχηθώ και καλή χρονιά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, διπλωμάτες, κυρίες και κύριοι. Και Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να πούμε ε, κάποια πράγματα για το σχέδιο δράσης της, προεδρίας, ε, της προσωρινής Προεδρίας της Κωνσταντίνας όσον αφορά το θέμα της ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Πριν ε, σας τα πω αυτά, να σας πω ότι θα αναφερθώ σε μια σειρά από δράσεις ε, και δραστηριότητες οι οποίες ως ε, σημείο αναφοράς ε, έχουν τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στη Μανάγκουα τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι ιδέες τις οποίες προτείνει η Κωνσταντίνα και ακόμα βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο, δεν έχουν εγκριθεί από όλε τι χώρε που συμμετέχουν στο σύστημα, βάσει των προθεσμιών του εσωτερικού κανονισμού. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, ε, επειδή υπάρχουν και κάποιες καινοτόμες ιδέες, ε, έχουμε κάνει επαφές ε, με την Δημοκρατία του Παναμά, η οποία θα αναλάβει την προσωρινή προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο, με στόχο να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και σχεδιασμός των δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, ε, η Κωνσταντίνα συνειδητοποιεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της έγκρισης, ένα στάδιο το οποίο ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2016 με μια συνεδρίαση ε, στην οποία συμμετείχαν διάφορες χώρες και η Γενική Γραμματεία και στις 19 Ιανουαρίου του 2017 έγινε η επόμενη συνεδρίαση. Ε, στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε το πλήρες πρόγραμμα ώστε να το χρησιμοποιήσουμε και να υπάρχει ως οριστικό κείμενο το οποίο θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Κατά, την άσκηση της Προεδρίας της η Κωνσταντίνα θα φροντίσει να ε, τηρηθούν και ε, ε, θα παρακολουθήσουμε και αυτή την τήρηση των ε, προεδρικών διαταγμάτων για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα εύρωστο, διάφανο πρόγραμμα με ε, κατάλληλες ηγετικές ικανότητες και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές προκλήσεις καθώς και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της περιοχής. Η δέσμευση της Κωνσταντίνας είναι να εργαστεί για την εφαρμογή και ενίσχυση του συστήματος σε θεσμικό επίπεδο ώστε να προχωρήσουμε σε θέματα διαφάνειας κυρίως και να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα που είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι η Ρίκα θα ε, ασχοληθεί με τις πέντε προτεραιότητες που ήδη έχουν ε, καθοριστεί για την ε, περιοχή. Δημοκρατική ασφάλεια, διαχείριση των κινδύνων της αλλαγής του κλίματος, ε, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας, κοινωνική, οικονομική ολοκλήρωση και ενίσχυση των θεσμών. θα έχουμε το θεματολόγιο του 2030 για την ανάπτυξη επίσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάθε προτεραιότητα θα την αντιμετωπίσουμε ε, μεμονωμένα, θα προτείνουμε συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες και, για παράδειγμα, όσον αφορά την ενίσχυση των θεσμών, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον κανονισμό εργασίας και της Προεδρίας, αλλά και να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό να υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία θα δίνονται λογαριασμοί, ε, θα γίνεται εξέταση των εντολών και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσουν η διαδικασία των διορισμών ε, των βασικών γραμματιών του συστήματος, κυρίως τη Γενική Γραμματεία του ΣΥΚΑ και τη Γραμματεία του Συστήματος Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Όσον αφορά το θεματολόγιο της οικονομικής ε, ένταξης ε, θέλουμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της ε, στρατηγικής της Κεντρικής Αμερικής για το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα, την πολιτική της κινητικότητας και του εφοδιασμού και ε, θέλουμε να έχουμε μια περιφερειακή έκθεση της κατάστασης των πολιτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα φόρουμ ε, δημοσίων συμβάσεων και τη στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, με γνώμονα την κεντροαμερικανική περιοχή. Θέλουμε επίση να προχωρήσουμε και τη Συμφωνία Σύνδεση Κεντρική Αμερική Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι ε, ακριβώς του συστήματος ΣΥΚΑ, αλλά ε, καλύπτει αρκετέ χώρες του συστήματος και γι' αυτό ακριβώ και ζητήσαμε να υπάρχει ε, εγκαίρωση, έγκριση από πλευρά κοινοβουλίων και επίση θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε και για τα όσα έκανε και η Πρόεδρο Σακοράφα αλλά και η αντιπροσωπεία σας ε, για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το ε, θεματολόγιο για την τουριστική ολοκλήρωση, θέλουμε να συνεργαστούμε σε διάφορα επίπεδα για να συμπεριλάβουμε και την συνιστόσα αυτή για την ε, στρατηγική της Κεντρικής Αμερικής για το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα, για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερο τουρισμό στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Όσον αφορά τη δημοκρατική διάσταση, θέλουμε να προχωρήσουμε τα θέματα της Επιτροπής Ασφαλείας και να εκτελέσουμε τα σχέδια εργασίας ε, της Υποεπιτροπής ε, και των συμφωνιών που έκαναν ο Υπουργό Εξωτερικών Ασφάλειας και Διακυβέρνησης που εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015 στο Σαν Σαλβαδόρ. Επιπλέον προτείνεται να οριστικοποιηθεί η αναθεώρηση του εσωτερικού ε, κανονισμού της Επιτροπής Ασφαλείας για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως οδικό χάρτη για να εκπονήσουμε ένα περιφερειακό σχέδιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, για να ε, πατάξουμε το έγκλημα με τη συμμετοχή των πολιτών. Όσον αφορά την κοινωνική ολοκλήρωση και την καταπολέμηση της ένδυας, κάποιες από τις ιδέες που προτείνονται είναι να υλοποιήσουμε προγράμματα και σχέδια που θέλουν να καταπολεμήσουν αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το δίκτυ της πολυδιάστατης ένδυας, ε, κοινωνικούς χάρτες και το σύστημα ε, διοργανικής συνεργασίας. Επίσης, θα υπάρχουν και κάποιες τεχνικοπολιτικές δραστηριότητες για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε επιτυχημένες εμπειρίες και να έχουμε δημόσιες πολιτικές. Όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του κλίματος, τέλος, ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει μια διάσκεψη για το νερό, για να μπορέσουμε να δούμε τι συνέπειες υπάρχουν λόγω της ξηρασίας στην περιοχή, καθώς επίσης και να οριστικοποιήσουμε την εκπόνηση ενός προγράμματος, το οποίο ε, ονομάζεται διάδρομος της ξηρασίας στην περιοχή και θέλουμε να δούμε πώς επηρεάζει η αλλαγή του κλίματος και να ολοκληρώσουμε την εντολή που... Ε, ε, εγκρίθηκε στην ε, ε, δήλωση. Όσον αφορά τις πολιτικές εκτός της περιφέρειας, ξέρετε ότι η ΣΥΚΑ διαθέτει αρκετούς παρατηρητές και μαζί τους θέλουν να κάνει εργαστήρια εργασίας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ε, περιοχές κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως για να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει πολιτική προσέγγιση, δυνατότητες εμπορίου και καθορισμός ε, μηχανισμών συνεργασίας, που θα είναι όλο ένα και πιο αποτελεσματική. Όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας, ε, τίθεται το θέμα της εφαρμογής του μηχανισμού διαχείρισης, συντονισμού και ε, ενημέρωσης ε, της ε, περιφερειακής συνεργασίας. Είναι περίπου 25 οι χώρες που συμμετέχουν ως παρατηρητές και στην Κεντρική Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα πολύ σημαντικό καθήκον που έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα είναι να υπάρχει ε, συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία και με τα Υπουργεία τα οποία ε, εκπροσωπούνται στο σύστημα με στόχο να ξεκινήσουν διαδικασίες διάρθρωσης σε όλα τα επίπεδα ε, και να υπάρχει και λογοδοσία η οποία θα υλοποιηθεί στις καθημερινές εργασίες της Γραμματείας. Τα όργανα τους, τα θεσμικά όργανα και τις χώρες οι οποίες ασκούν την προσωρινή Προεδρία. Τέλος, ε, για την Κωνσταντίνα, ε, μας ενδιαφέρει το ίδιο πρωτόκολλο της Κουσιγάλπα που στο άρθρο 3 προβλέπει ότι το βασικό είναι να υπάρχει μια περιοχή ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας και ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, είμαι και εγώ σίγουρη ότι θα αναλάβετε όλε εκείνε τι θεσμικέ πρωτοβουλίε ώστε να αντιμετωπίσετε όλε τι προκλήσει πολιτικέ, οικονομικέ, τι οποίε έχετε μπροστά σα και θα αντιμετωπίσετε. Ε, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντελαρίτσια, ε, επικεφαλή του τμήματο για την Κεντρική Αμερική, Μεξικό και Καραϊβική από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Κύριε Ντελαρίτσια, έχετε το λόγο. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Señores diputados, Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μακρά ιστορία ε, σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, μια μακρά ιστορία εταιρική σχέσης ε, που βασίζεται στην κοινή δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε υποστηρίξει τη ΣΥΚΑ, τους θεσμούς της ε, που είναι στη βάση αυτής της προσπάθειας ολοκλήρωσης της ε, περιοχής της Κεντρικής Αμερικής. Η ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής είναι ένα σημείο κλειδί για τη σταθερότητα αλλά και την ευημερία της περιοχής. Όλε, ε, όλες οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή, η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ολοκλήρωση, η συνοχή, ή το διασυνοριακό έγκλημα ή μετανάστευση, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να τα αντιμετωπίσει κανείς καλύτερα από κοινού, σε περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ακούμε αυτά που προετοιμάζει η Κωνσταντίνα για αυτήν την προσωρινή προεδρία και καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της ΣΥΚΑ να ε, συνεργαστούν, να συνεισφέρουν σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει μια κοινή ατζέντα μεταξύ Κωνσταντρίκας και, και Παναμά. Είναι πολύ επικοδομητική αυτή η ιδέα, μιας και η συνοχή καθώς και η συνέχεια καθιστούν πιο αποτελεσματική την όλη προσπάθεια, την όλη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης. Υποστηρίζουμε επίσης ε, όλη την ατζέντα θεσμικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής του Ουατάν και επικυρώθηκε στη Μανάγκουα. Θα θέλαμε επίσης να υπογραμμίσουμε τη σημασία της συνένεσης στα πλαίσια του συστήματος ε, ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υποστηριχθούν από, από όλους. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Κοσταρίκα σε αυτή την κοινή δράση με τον Παναμά ε, θα λάβει υπόψη αυτήν την πτυχή της αρμονίας. Το 2017 θα υπάρξει μια αλλαγή πλεύσης στην ΣΥΚΑ ε, αλλά και στις διευθύνσεις της. Ε, εμείς είμαστε πάρα διατεθειμένοι βέβαια να υποστηρίξουμε τη ΣΥΚΑ στη διαδικασία αυτή καθώς και την Κοσταρίκα ως προσωρινή προεδρία της ΣΥΚΑ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως περνάει και αυτή τη δική της κρίση. Έχουμε κι εμείς ε, μια κάποια εμπειρία την οποία μπορούμε να μοιραστούμε με την Κεντρική Αμερική. Θα ήθελα με την ευκαιρία να, υποστηρίξω, να υπογραμμίσω συγγνώμη, τη σημασία της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ως βασικό εργαλείο στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Αμερική. Υπάρχει συμφωνία σύνδεσης η οποία έχει να κάνει με το εμπορικό σκέλος και υπάρχει και συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, πολύ σημαντικό στοιχείο ε, μια συνεδρία που εκρεμεί από πέρσι, καλό θα ήταν να λάβει η χώρα έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στη συνεργασία με την Κεντρική Αμερική. Την περίοδο 2014-2020 είχαμε μια σημαντική αύξηση της συνεργασίας για το σύνολο της περιοχής αυτής. Μιλάμε για 925 εκατομμύρια ευρώ και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της υποπεριφερειακής ε, συνεργασίας από αυτά τα 925 εκατομμύρια έχουν διαιρεθεί 120 για αυτή τη διαδικασία. Ένα από τα παραδείγματα του πώς αυτή η συνεργασία εκτελείται, λαμβάνει χώρα, έχει να κάνει με την, την υποστήριξη του κρίσιμου τομέα ε, της ασφάλειας των πολιτών. Μπορέσαμε έτσι να εφαρμόσουμε ε, αυτή τη στρατηγική υποστήριξης Τη ασφάλεια των πολιτών στην Κεντρική Αμερική και στην Καραϊβική ουσιαστικά ερχόμαστε να υποστηρίξουμε στρατηγικέ που υπάρχουν ήδη στην περιοχή και είναι σημαντικό το ότι η Προεδρία, η προσωρινή Προεδρία τη Κωνσταντίνα, ε, δίνει προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Νταρέτσια, τώρα το λόγο έχουν τα μέλη μας. Ε, έχω γράψει την κυρία Γιούζο, ζήτησε το λόγο, ο κύριος Φαρία μετά. Δεν ξέρω κάποιος άλλος, κυρία Τσίνηση. Θέλετε το λόγο και εσείς. Η κυρία Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους πρέσβεις ε, και τους υπολείπους ε, προσκεκλημένους, τον επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικής Δράσης και επίσης να σας πω ότι όλο σας το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ φιλόδοξο σίγουρα μπορεί να υλοποιηθεί και σας εύχομαι και εξαιρετική προσωρινή προεδρία. Ήθελα ε, να μιλήσω για την πρώτη σας παρέμβαση, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το ταξίδι που μας ανακοινώσατε ε, για την Κούβα. Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικό να υπάρχει αντιπροσωπεία στην Κούβα, διότι έχουν ξεκινήσει και κάποιες αλλαγές στις σχέσεις, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω ε, προηγουμένως να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία στις επαφές που θα κάνουμε στο ταξίδι αυτό, ελεύθερη κυκλοφορία και ελευθερία κινήσεων εντό του νησιού. Ε, πριν δεσμευτούμε για αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα τηρηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όσα ταξίδια τουλάχιστον έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, στις χώρες που έχουμε επισκεφθεί, δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ τέτοιου είδους πρόβλημα. Και πιστεύω ότι και στην επίσκεψή μας, εάν ευοδοθεί στην Κούβα, θα είναι ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Ο κύριος Φαρία έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω και εγώ τον πρέσβη. Ε, δεν πρόλαβα όλη την ομιλία σας γιατί καθυστέρησα. Ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξή όσον αφορά την Προεδρία στην ΣΥΚΑ, στο Σύστημα Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Θέλετε να προωθηθεί η ολοκλήρωση στην Κεντρική Αμερική και θέλω να σας ρωτήσω Πώς βλέπετε την νέα Αμερικανική διοίκηση και τις ε, απομονωτικές της απόψεις, ειδικότερα όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής. Είχαμε την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε το, από το 1991. Ε, τι πρόκειται να συμβεί κατά την άποψή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Κίνητση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη διοργανώση αυτής της συνάντησης ε, της αντιπροσωπείας μας και ευχαριστώ τους πρέσβεις και όλους τους ε, καλεσμένους. Συμφωνώ με τα εισαγωγικά λόγια της Προέδρου ότι οι περιοχές για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ε, αναταράξεις και καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές προκλήσεις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές. Εκτίμησα ιδιαίτερα όσα υπόθηκαν ε, είτε από τον πρέσβη Αλφαρό όπως και από τον ε, κύριο Ντελαρίτσα όσον αφορά τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί. Στόχοι φιλόδοξοι πρέπει να πω, σύμφωνα με τους οποίους φυσικά εμείς ευχόμαστε να επιτευχθούν όλοι και πιστεύουμε ότι συνεχίζοντας τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα ακούγοντας ε, την παρουσίαση των στόχων αυτών. Επισημένοντα ορισμένου, ορισμένους μόνο, ε, γιατί είναι ιδιαίτερα ευρύς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αλληλένδετη. Γιατί όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, την ασφάλεια κτλ. Δύο ερωτήσεις λοιπόν ε, ή μάλλον ε, ζητώ δύο διευκρινήσεις, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εντός της αντιπροσωπείας, εγώ δεσμεύομαι πολιτικά πάρα πολύ στα, ως στα ανήλικα παιδιά και είμαι πεπισμένη ότι τόσο στις περιοχές της Κεντρικής Αμερικής όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυση στους νέους σημαίνει επένδυση στο εγγύς μέλλον των χωρών μας. Συνεπώ ε, πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης των κοινωνικών συνθήκων, οικονομικών, των δικαιωμάτων, των συνθήκων ασφαλείας, ειδικότερα όσον αφορά τους νότερους. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχουμε πολλούς, πολύ αριθμούς στόχου, πολύ φιλόδοξου, και εύχομαι να του επιτύχουμε. Αλλά έχουν προβλεφθεί κάποιε προτεραιότητε. έχουμε σκεφτεί υπό ποιε προποθέσει θα επενδύσουμε στου νεότερους αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχόμενη επαναλαμβάνω να μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση επιτυχώς και να βελτιώσουμε τα πράγματα επιτυγχάνοντα όλους τους ε, στόχου που έχουμε προκαθορίσει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρεσβή, ο λόγο είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση, η Κεντρική Αμερική έχει μια συμφωνία ολοκλήρωσης ε, η οποία είναι ανεξάρτητη και το πρωτόκολλο για το 91 ε, μας επιτρέπει να μπορούμε να κάνουμε κοινέ δράσεις ε, σε μια περιοχή που είναι η άμεση περιοχή μας, η άμεση γειτονία μας. Επομένως θεωρείται εσωτερικό θέμα αυτό. Θεωρώ ότι όλες οι χώρες ε, της περιοχής κάνουν το ίδιο, αλλά στην περίπτωση της Κωνσταντίνας η καλύτερη λύση είναι να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, γιατί στην αρχή της αλλαγής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ε, μας δείχνουν ε, και κάποιες αλλαγές ε, οι οποίες γίνονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πράγματι, ε, στην περίπτωση της ε, θα πρέπει να συντονίσουμε την σύνοδο στο Γουτέρες και θα περιλαμβάνεται και το Μεξικό και υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις που αφορούν τις εσωτερικές σχέσεις Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς θα κάνουμε ανάλυση, αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τα διάφορα ενδεχόμενα και θα δούμε αν κάποια στιγμή η περιοχή ε, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη και επομένως ε, προσέχουμε απλώς ε, την κατάσταση. Όσον αφορά τα όσα ανέφερε η κυρία Κινίτση για την παιδική ηλικία και την, βρεφική, και την εφηβική ηλικία, η Κώστα Ρίκα από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχουμε υπογράψει. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική δουλειά για να μην υπάρχει παιδική εργασία, να υπάρχουν ε, ε, δημόσιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα προωθούν περισσότερο την εκπαίδευση ε, και από την εργασία και βεβαίως η χώρα πρέπει να σεβαστεί και κάθε ένα από τα εσωτερικά συστήματα στις υπόλοιπες χώρες. Βεβαίως, επίσης, ε, υπάρχουν και μία σειρά από δράσεις τις οποίες αναφέρατε, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες. Ε, θα μπορούσαμε να σας δώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ήδη εγκρίνει, όταν ε, όλες οι χώρες θα μπορέσουν να συμμετέχουν και θα μπορέσουν να δουν και όλες οι δράσεις πώς υλοποιούνται. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις απεξηγήσεις που μας δώσατε. Και τώρα θα πρέπει να πάμε στο έκτο σημείο της σημερινής ε, ημερήσιας διάταξής μας που αφορά στην έκθεση νούμερο 30 κάθετος 2016 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα. Το ζήτημα τη στήριξη, κύριε συνάδελφοι, και τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κεντρική σημασία για τι σχέσει των χωρών τη Κεντρική Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση η φύση αυτή τη στήριξη αλλάζει δραματικά και ω εκ τούτου είναι χρήσιμο να γίνει ένα απολογισμό τη αποτελεσματικότητα τη στήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν. Υπό αυτή την έννοια χαιρετίζω θερμά τη δημοσίευση τη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα τη στήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομεί προτεραιότητα στην Ονδούρα και είμαι πεπισμένη ότι οι διαπιστώσει των ελεγκτών θα μα διδάξουν σημαντικά μαθήματα και το πώς να σχεδιάσουμε καλύτερα τις μελλοντικέ πολιτικές συνεργασίες προς αμοιβαίο όφελος βεβαίως των χωρών της Κεντρικής Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα εδώ να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάκομσεν, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να μας πει τα της έκθεσης. Κυρία Γιάκομσεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτοεξοχότητες, ε, μέλη της αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Λατινική Αμερική, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για την αποτελεσματικότητα της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα. Στα αριστερά μου να σας παρουσιάσω τον επικεφαλής ε, των εργασιών αυτών, τον κύριο Βλασλάρ, ε, στην παρουσίασή μου θα παρουσιάσω συνοπτικά τα κυρία ευρήματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Αλλά πρώτα να σας ε, δείξω ποια είναι η γενική εικόνα της ευρωπαϊκής υποστηρίξης προς την Ονδούρα. Χώρα που έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, ε, υποφέρει από μεγάλη φτώχεια, αστάθεια, πολιτική, βία, και άλλα προβλήματα. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός ε, εταίρος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ονδούρας ε, και ο μεγαλύτερος δωρετής. Το κονδύλιο από 223 εκατομμύρια ευρώ το 2007 έχει πάει στα 2,35 εκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020. Για την περίοδο που εμείς ελέγξαμε στην έκθεση μας από το 2007 μέχρι το 2015 οι πληρωμές ανέρχονταν σε 190 ε, εκατομμύρια ευρώ με σχεδόν μισή από τη διμερή η στήριξη να παρέχεται ως στήριξη του προπολογισμού και το άλλο μισό υπό τη μορφή έργων. Πέραν αυτών, η Ονδούρα επίσης επωφελήθηκε από περιφερειακά, ε, προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, υποπεριφερειακά προγράμματα και θεματικές γραμμές του προπολογισμού. Στον έλεγχο μας εξετάσαμε τους τρεις τομείς προτεραιότητας, ε, μείωση της φτώχειας, φυσική πόρη και ασφάλεια και δικαιοσύνη, που έλαβαν όλοι μαζί το 89% των δαπανών της δημερού Ο έλεγχος μας ε, αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα. Πραγματοποιήσαμε την αξιολόγηση ε, εξετάζοντας πρώτα απ' όλα τη διχείριση εκ μέρους της ε, Επιτροπής ε, της Αναπτυξιακής Στήριξης και δεύτερον ε, τον βαθμό επίτευξης των στόχων. Ποια ήταν τα ευρήματα. Συνολικά το μήνυμα της έκθεσης είναι ότι η διμερής αναπτυξιακή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στην Ονδούρα κατά την περίοδο ελεγχού ήταν μερικώς αποτελεσματική. Στις δύσκολε συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα, οι δράσει τη Ευρωπαϊκής Ένωση έκαναν μια διαφορά και γενικά παρήχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρότι ενίοτε με καθυστερήσει και η στήριξη συνέβαλε σε μια σειρά θετικών εξελίξεων. Από την άλλη πλευρά, η γενικότερη κατάσταση της χώρας παραμένει ενισχυτική. Το επίπεδο της φτώχειας έχει αυξηθεί ε, οι δασικές περιοχές ε, έχουν μειωθεί σε έκταση και υπάρχει ευρεία βία και πολύ ψηλό ποσοστό ανθρωποκτονιών. Επίσης ε, ανακαλύψαμε αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης της ευρωπαϊκής αρρωγής από τις Κομισιόν. Παρότι η προσέγγιση της Επιτροπής για την παροχή αναπτυξιακής στήριξης στην Ονδούρα στόχευσε σωστά τομείς υψηλής ανάγκης, που καλύπτονται από εθνικές ε, στρατηγικές ε, παρουσιάστηκαν σημαντικές ελλείψεις. Η ευελιξία της προσέγγισης της Επιτροπής ε, σήμανε ότι ορισμένοι τομείς έλαβαν ευρωπαϊκή στήριξη για σχετικά μικρό διάστημα. Γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο να μην επιτευχθούν τα αποτελέσματα που, είχαμε επιθυμεί, που επιθυμούσαμε. Επίσης, η επίδειξη των στόχων και η οικονομική βοήθεια μοιράστηκε σε πολλού τομεί. Παρότι υπάρχει σωστό συντονισμό μεταξύ των δωρετών στην Ονδούρα, η πραγματική συνεργασία ήταν κάτι σχετικά περιορισμένο. Γεγονό που δείξε σε επικαλύψει τη στήριξη σε ορισμένε περιπτώσει. Η υποστήριξη του προπολογισμού στην Ονδούρα ήταν κάτι επικίνδυνο λόγω του ασταθού μακροοικονομικού πλαισίου και της αδύναμης ε, ε, διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Παρότι η Επιτροπή κατάφερε να μετριάσει τους κίνδυνους αυτούς σε κάποιο βαθμό, δεν αξιολόγησε την επιλεξιμότητα της στήριξης ε, του προπολογισμού με αρκετά δομημένο τρόπο για να δείξει ότι η πρόοδος της χώρας ευθυγραμμιζόταν με συγκεκριμένους στόχους και benchmarks. Οι περισσότερε προγραμματισμένε δραστηριότητε και τα περισσότερα προγραμματισμένα αποτελέσματα επιτεύχθησαν, αλλά με καθυστερήσει κυρίως λόγω εξωτερικών παραγόντων. Η παρακολούθηση επιδόσεων της Επιτροπής επηρεάστηκε από δυναμία επιλογής ε, και χρήσης δικτών ε, και από δυναμίες στο follow-up των συστάσεων. Η Επιτροπή ανέπτυξε στρατηγικές ε, για επικοδομητικό πολιτικό διάλογο σε διάφορους τομείς με την κυβέρνηση της Ονδούρας Παρότι η πρακτική αυτή είναι καλή, αυτοί οι στρατηγικέ επιτροπέ ε, τείνουν να είναι γενικολογέ και όχι να καλύπτουν όλου του ε, ε, σημαντικού τομεί. Τι συνιστά λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο? Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της στήριξης Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τη συνοχή και την εστίαση. Συνιστούμε λοιπόν η Επιτροπή να ενισχύσει τέσσερι τομεί. Ο πρώτο είναι η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύοντας την εστίαση και τη συνοχή. Δεύτερη είναι η διαχείριση τη δημοσιονομική ε, στήριξη ε, και των σχετικών δράσεων. Τρίτον, ε, μέτρηση επιδόσεων των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και τέλο διάλογο πολιτική στους τομεί προτεραιότητα. Επιπροσθέτω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την επικοδομητική του συνεργασία κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού και για τη δέσμευση που έδειξε αποδεχόμενοι όλες τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για την επιδείξη περαιτέρω βελτιώσεων στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήσει που ενδεχομένως έχετε για την έκθεση ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα να δώσω τον λόγο στον, στην αυτοεξοχότητα των πρέσβη, τον κύριο Τσόμαντρη, πρέσβη της Ονδούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο.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 que incorpora periodos gubernamentales de crisis política, establecimiento democrático, unidad nacional. Υπήρξαν πολιτικές κρίσεις, υπήρξαν μεταρρυθμίσεις, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση του Τσοντούρας ε, χαίρεται που έχουμε λάβει χώρα όλες αυτές τις δραστηριότητε ε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτές τις, ε, αυτή την ενίσχυση. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Ε, σε αυτή την περίοδο υπήρξε μια έρευνα παρακολούθησης του Παρισιού και υπήρξε επίσης μια έκθεση για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης και βεβαίως η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πιο σημαντική ε, για τη χώρα μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχει να, κάνει, έχει να κάνει με την ε, εξοικείωση και την οικειοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν ο διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης της Ονδούρας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρούμε και άλλες κοινέ δράσεις για να υπάρξει μια βελτίωση ε, των της, της συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί και ο διάλογος του τομεί προτεραιότητας πριν από το 2018. Ε, θα πρέπει να δοθεί μια νέα δυναμική στη στρατηγική ε, για την παρακολούθηση των διαφορών σχεδίων. Υπάρχουν προτεραιότητες ό,τι αφορά τις ζώνες παρέμβασης βέβαια. Ε, εμείς ε, θα θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την ε, Επιτροπή Παρατηρητών ε, Εκλογών τα τελευταία χρόνια. Οι δύο τελευταίες εκλογές ε, ήταν και πλέον δημοκρατικές και με σπέστος παρατηρητές τα σχόλια των παρατηρητών της Ευρώπης μας οδήγησαν στο να μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε το εκλογικό συμβούλιο αλλά και το εκλογικό νόμο καθώς και τον νόμο χρηματοδότησης ε, της προεκλογικής εκστρατείας για, που έχει οδηγήσει μεγαλύτερη διαφάνεια τα πολιετή, τα προγράμματα και η, επιλογή των τομέων υποστήριξης έγινε με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο προϋπολογισμός για το 2013 έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση ε, για σχέδια τα οποία έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ε, έχουμε λάβει υπόψη τις προτεραιότητες της δικής μας κυβέρνησης βέβαια. Ε, υπάρχει το θέμα της δημοσιονομικής υποστήριξης που έχει την υποστήριξη τα εθνικά συστήματα. Προσπαθούμε να υπάρχει μια προλεψιμότητα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση. Θέλουμε μια στρατηγική μακροπρόθεσμη εξαετή που δίνει τη δυνατότητα στην Ονδούρα να προετοιμάσει καλύτερα τα προγράμματα συμπληρώνοντας ε, και σε εθνικό επίπεδο τη χρηματοδότηση σε διάφορε τομεί, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη, ασφάλεια. Χάρη στην υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα προχώρησε. Προχώρησε, ε, σημείωσε σημαντική πρόοδο. Έχουμε ενισχύσει του θεσμού, του δικαστικού μέσω του προγράμματο Euro για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, την εγκληματικότητα και να, έχουμε, να υπάρχει μια πρόσβαση σε ένα δικαστικό σύστημα γρήγορο, αποτελεσματικό και ισότιμο. Χάρη στην συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ενισχύσει επίσης τη δημιουργία της αποστολής ε, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ε, τα μέσα που μας παρέχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε θεσμικό, σε θεσμικό επίπεδο να μπορέσουμε να πολεμήσουμε τη διαφθορά και την ατιμορρησία η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άλλων φορέων μας έχει οδηγήσει ε, στο να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο ε, της εξυγίανσης και των αστυνομικών μας αρχών, των αστυνομικών δυνάμεων, έτσι ώστε η αστυνομία μας να οδηγήσει η ίδια σε σημαντικές αλλαγές. Έχουμε αντιμετωπίσει βεβαίω σημαντικές δυσκολίες. Είχαμε 25 επιχειρησιακά σχέδια ε, ε, χάρη στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον δασικό τομέα επίσης έχει υπάρξει δημοσιονομική υποστήριξη για την ταυτοποίηση των περιοχών που θα πρέπει, όπου θα πρέπει να υπάρξει αναδάσωση για την προστασία των φυσικών πόρων γενικότερα. Έχουν προχωρήσει διαπραγματεύσει σύνδεσης και αυτό συνοδεύεται από μια διαβούλευση που σέβεται ε, τις αρχές ε, της ε, ε και πρώτερης ε, συμμετοχής οργανώσεων περιβαλλοντικών με την, την υπογραφή του ΑΒΑΦΛΕΤ εμείς είμαστε είμαστε πρώτη χώρα που θα μπορεί να εξάγει ξυλία πιστοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε φτάσει σε συμφωνία και με το Διεθνές Ομοσπονδικό Ταμείο πληρών, εφόσον πληρούμε βέβαια τις ε, ε, συμβουλές τους, ε, υπάρχουν διάφοροι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ε, και δημιουργείται ένα κλίμα πιο κατάλληλο ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην δημοσιονομική υποστήριξη. Ε, το ίδιο το Ταμείο αναφέρεται στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3,6% πέρυσι και ο στόχος για φέτος είναι 3,7%. Ε, υπάρχει λοιπόν μια μακροοικονομική σταθερότητα στη χώρα μας που μας επιτρέπει να ε, προβούμε σε αυτή τη δημοσιονομική υποστήριξη. Ε, στην Ονδούρα και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της μείωσης της φτώχειας. Βεβαίως δεν έχουμε επιλύσει όλα τα δύσκολα ζητήματα, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία μας αντιμετωπίσαμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά, το εμπόριο ναρκωτικών, ε, τις διάφορες πύρες ε, και, και αυτό έγινε με συστηματικό και μόνιμο τρόπο. Υπάρχει πολιτική βούληση και του λαού και της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κακά. Είμαστε βέβαιοι ότι στην επόμενη περίοδο ελέγχου του Λετικού Συνεδρίου θα φανούν ακόμα περισσότερο αυτά τα βήματα πρόοδου σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, ε, μάλλον χάρη και στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρέσβη, να δώσω το λόγο στην κυρία Μπούτκε Βιέντσε, προϊσταμένη της Μονάδας για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη. Um, thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τους μεταφραστές, για τους διερμηνές. Ε, το όνομά μου είναι Γιολίτα. Αλλά δεν πειράζει που το είπατε λάθος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω τις εντυπώσεις μου από το μέρος το ίδιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρέζιο για την πολύ πιστική σας δήλωση όπου ε, στην ιστοσελίδα που αναγνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση Ω εταίρο. Μακάρι να μπορούσαμε να εργαστούμε όλοι στην Κωνσταντίνα μόνο, αλλά έχουμε πολλές χώρες στην Λατινική Αμερική και έχει αναγνωριστεί ήδη ότι έχουμε πολλή δουλειά και στην Ονδούρα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει μια κυβέρνηση μέσα σε μια τετραετία. Η κατάσταση οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες όπως έχει αναγνωρίσει το Ελληνικό συνέδριο. δεν είναι πλέον η χώρα με τις περισσότερες ανθρωποκτονίες και το λέω με ευχαρίστηση. Αλλά η ζωή στην Ονδούρα και η δουλειά στην Ονδούρα δεν είναι κάτι εύκολο η καθημερινότητα. Τώρα, αν δείτε ε, το κονδύλιο που είχαμε πάνω από 200 εκατομμύριο ευρώ με τη δική σας, συμφωνία για τη χώρα αυτή των 8 εκατομμυρίων, ε, αυτό το ποσό μας περιορίζει στο τι μπορούμε να επιτύχουμε. Δεν μπορούμε πραγματικά να πολεμήσουμε τη φτώχεια. Μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να πολεμήσει τη φτώχεια. Το διάστημα που καλύφθηκε, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από το Ελληνικτικό συνέδριο, κάλυψε τεράστιους ε, τομείς, τεράστιες περιοχές, γιατί η βασική μας εστίαση ήταν να υποστηρίξουμε το εθνικό σχέδιο της Ονδούρας για την αντιμετώπιση της φτώχειας, κάτι που συνεπάγεται πολλές κοινωνικές υπηρεσίες. Ε, περιλαμβάνει πολλές κοινωνικές υπηρεσίες και αυτό φαίνεται έτσι πολύ ευρύ. Αλλά ε, το 2007 ξεκινήσαμε και στο μεταξύ γίναμε πιο σαφή, πιο σοφή, πιο αυστηρή με τις ε, δράσεις μας και έτσι εστιαστήκαμε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και υποστηρίξαμε τις περιοχές και τους τομείς που, στους οποίους είχε προτεραιότητα η κυβέρνηση εκείνη την εποχή. Γι' αυτό το λόγο το ελεγκτικό συνέδριο βλέπει ελλειπή εστίαση και διάχυση σε πολλούς τομείς. Οι αλλαγές που συνέβησαν ήταν αυτές που ανέφερε ο πρέσβης ακριβώς εμείς είμαστε γνωστοί και ως ευέλικτος εταίρος. Ανταποκρινόμαστε σε επίρουσες ανάγκες ε, και όταν υπήρξε ε, πραξικόπημα χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση και στις δράσεις που θα υποστηρίζαμε επί τόπου. Φυσικά στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, το οποίο ήδη καλύψατε, ε, η εστίαση είχε περιοριστεί, οι τομεί δηλαδή με του οποίου ασχοληθήκαμε σε συμφωνία με την κυβέρνηση ήταν πιο εστιασμένοι. Δεν ε, αντιμετωπίζαμε την φτώχεια γενικότερα, αλλά τη διατροφική ασφάλεια, την απασχόληση, κάτι που καλυπτόταν από, μια, από την ενιαία ε, γενική προσέγγιση. Και έτσι εξελίχθηκε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα και τη εξέλιξη του τρόπου που εμεί σκεφτόμαστε και των πρακτικών που εφαρμόζουμε, ε, ώστε να φέρουμε κάπω καλύτερα, παραπάνω αποτελέσματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερου που εργαζόμαστε στην Ονδούρα για πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα, διότι έχουμε δέσμευση τη κυβέρνηση να συνεργαστεί μαζί μα. Όπω αναγνωρίζει, πιστεύω και το ελεκτικό συνέδριο ω Ευρωπαίοι, μπορούμε να είμαστε ε, περήφανοι για το έργο που έχει επιτελεστεί στην Ονδούρα, διότι πρόκειται για χρήματα που επενδύθηκαν για πραγματική υποστήριξη τη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα ε, ευρωπαϊκά χρήματα που μπαίνουν στη χώρα και οι πόροι συγκριτικά είναι πολύ μικροί αν τους συγκρινούμε με το τι έχουμε επενδύσει σε άλλες ε, χώρες. Είμαι επίσης ειδικότερα περήφανη για το συντονισμό των δωρητών. Φυσικά, αν δει κανείς απομονωμένα την Ονδούρα, παρατηρεί ε, κάποιες επικαλύψει. Όλοι πάμε στις ίδιου τομεί, στους ίδιου Δήμου, ε, για να εργαστούμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους, ε, διότι είναι πολιτικά σημαντικές, αλλά και γιατί είναι περιοχές όπου πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η, η περιοχή του, του ξηρού διαδρόμου που είναι γνωστή για τα θέματα διατροφικής ασφάλειας ήταν ένας τομέας στον οποίο εστιαστήκαμε και πετύχαμε πολλά. Είχαμε την ομάδα των δωρητών που ονομάζεται Group 16, ένα από τα παραδείγματα ε, συντονισμού μας στη χώρα και το πώς ε, η ισχυρή οικειοποίηση από πλευράς κυβέρνησης βοήθησε στη συνεργασία με τους δωρητές. Όχι σε όλη την Λατινική Αμερική, αλλά σε ορισμένες χώρες κάποιες κυβερνήσεις προτιμούν να μιλάνε με συγκεκριμένους δωρητές, γεγονός που είναι κάποιο πλεονέκτημα. Αυτό δεν συνέβη στην Ονδούρα. Όταν αντιμετώπισε προβλήματα κάποια στιγμή η κυβέρνηση με τα διεθνή χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα, ο πρόεδρο κάθισε με την ομάδα των δωρετών, του εξήγησε την προσέγγιση πώ σκέφτεται να αντιμετωπίσει με την κυβέρνηση τα προβλήματα. Συγκριτικά λοιπόν με άλλε ώρε η Ονδούρα είναι υποδειγματική, θα έλεγα, ε, σε θέματα συντονισμού μεταξύ των δωρετών. Ε, συμφωνώ με το ελεκτικό συνέδριο δεν διαφωνώ με τίποτα. Απλά να πω ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο ακούγονται και ένα γενικό συμπέρασμα, στο γενικό συμπέρασμα το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει ότι δεν σπαταλήσαμε χρήματα, δεν χάσαμε τα χρήματα μας εκεί. Πρόκειται μια καλή επένδυση. Τώρα, αν ήταν η καλύτερη, θεωρούμε ότι δεδομένων των συνθηκών, ναι, ήταν. Τώρα, ένα τομέα περίπλοκο όπω η δικαιοσύνη και η ασφάλεια ε, συνεπάγεται την απέτηση εκπαίδευση πολλών ανθρώπων και πολλοί δωρητέ ε, ε, το έκαναν αυτό, πολύ χορηγοί. Το γεγονό ότι πολλοί κόσμος δούλεψε στη χώρα αυτή για την εκπαίδευση των αστυνομικών δεν σημαίνει ότι καλύψαμε τι ανάγκε τη χώρα. Οι προκλήσει είναι τόσο μεγάλε που όλοι οι χορηγοί μαζί και όλοι οι πόροι που έχει η κυβέρνηση, ακόμη και αν διατεθούν, όλοι οι πόροι που έχει στη διάθεσή τη η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βοηθήσουν να υπερβούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, διότι τα προβλήματα προέρχονται εκτός από τη, έξω από τη χώρα. Ε, και μια χώρα 8 εκατομμυρίων δεν έχει τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει. Εμεί φυσικά επίση. Ε, ε, μας απασχόλησαν ιδιαίτερα τα θέματα για τη δημοσιονομική διαχείριση ε, το Ελεκτικό συνέδριο και παλιότερα με τη γενική αξιολόγηση της δημοσιονομικής υποστήριξης και κοιτώντας πώς τη διαχειριστήκαμε το 2007 και πώς τη διαχειριζόμαστε σήμερα, πρόκειται για μέρα και τη νύχτα. Έχουμε μια πιο δομημένη προσέγγιση, πιο επικεντρωμένη ε, σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. Κάπου έχουμε τυποποιήσει πλέον τη δομή και βάσει των όσων όλα αυτά που συνιστά το ελεκτικό συνέδριο τα έχουμε ήδη υλοποιήσει πιστεύω σήμερα. Δηλαδή έχουμε ανταποκριθεί θα έλεγα αρκετά αποτελεσματικά στις συστάσεις του και παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Τώρα όσον αφορά τη διαχείριση της δημοσιονομικής στήριξης, και δεν μιλάω τώρα για τον εαυτό μου, μιλάω για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, των δράσεων. Χρειαζόμαστε ειδικού που να μπορούν πραγματικά να αξιολογήσουν την καθημερινότητα στη χώρα και αυτό ανέφερε το ελεκτικό συνέδριο Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εύκολο να προσλάβει κανείς ε, ε, ότι είναι δύσκολο να προσλάβει κανείς ανθρώπους για να πάνε να δουλέψουν στην Ονδούρα. Αν είχε κανείς την επιλογή μεταξύ Κωνσταντίνα και Ονδούρα, Ονδούρα θα πήγαινε κανεί στην Κωνσταντίνα και λυπάμαι που το λέω κύριε Πρέσβη. Είναι δύσκολη η κατάσταση στη χώρα και το σύστημα που έχουμε εμεί, το σύστημα πρόσληψη ανθρώπων, όλα τα συστήματα τη Επιτροπή έχουν διαφορού ενσωματωμένου ελέγχου, δεν είναι πολύ ευέλικτα. Και ξέρετε, ε, το να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο και την κατάλληλη θέση δεν είναι κάτι εύκολο. Απαιτείται χρόνος. Και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και να διαβεβαιώσω το ελεκτικό συνέδριο ότι εισάκουσε ο γενικός μας διευθυντής τη παρατηρήση σα και άρχισε αναθεώρηση ε, ε, όλων των αντιπροσωπιών για να είμαστε βέβαιοι ότι βρίσκονται κατάλληλα άτομα στι σωστέ θέσει και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους αλλά φυσικά υπάρχουν διάφοροι παράγοντες υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, μια από τι καλύτερε που υπάρχουν για την υποστήριξη τη δημοσιονομική διαχείριση προ την κυβέρνηση και τη μακροοικονομική διαχείριση επίση. Ε, εργαστήκαμε ε, πολύ στενά με το Δονοτού, με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είχαμε μεγάλη υποστήριξη ε, από το κέντρο και είχαμε και ανθρώπους που πήγαν για να υποστηρίξουν το προσωπικό μας εκεί. Παρότι λοιπόν η εμπειρογνωμοσύνη που προφέραμε δεν ήταν πάντα, ε, δεν ευθυγραμμιζόταν πάντα ακριβώ με ό,τι προσπαθούσαμε να πετύχουμε, ε, χρησιμοποίησαμε ε, διασφαλίσει ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση ε, σημείωσε πρόοδο σε κάποιου τομεί με τους δείκτες. Ξέρετε υπάρχουν κάποια όρια πρέπει να δει κανείς ποια είναι η βασική κατάσταση, επί το τα στατιστικά στοιχεία και βάσει αυτών ε, καθορίζει, τι θα, με, καθορίζει κανείς τι θα μετρήσει και πώς θα εκταμιεύσει κονδύλια ανάλογα. Όταν λοιπόν το, το στατιστικό σύστημα είναι ελλειπές, ε, Παρ' όλα αυτά, εμεί πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο το ελεγκτικό συνέδριο ανέφερε ότι οι δείκτε δεν ήταν απαραίτητα αξιόπιστοι σε όλε τι περιπτώσει. Με το οποίο συμφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρά ό,τι έχουμε στα χέρια μα. Και εμεί αυτό που υποστηρίξαμε ω προσέγγιση είναι ότι θα υποστηρίξουμε την πρόοδο. Ότι μαζί όλοι θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε προ ένα μελλοντικό στόχο και όλε οι επενδύσει μα γίναν βάση πρόοδου όσον αφορά τη φορολογική συμμόρφωση, αυξήθηκαν οι ελέγχοι ε, εντάθηκαν οι, τα πρόστιμα φοροδιαφυγής, ε, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ε, και με τους ε, σχετικούς φορολογικούς εισαγγελείς και τα λοιπά και θεσμοθετήθηκαν ειδικοί δικαστές για τα φορολογικά εγκλήματα σε όλη τη χώρα. Έγιναν λοιπόν κάποιες σημαντικές θετικές πρόοδοι. Μπορεί να μην αναφέρονται έτσι ρητά στους δείκτες, αλλά έχουμε επιτύχει και τη δέσμευση τη κυβέρνηση για να κινηθούμε προς τα εμπρός και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για ένα πράγμα ότι έχουμε μπροστά μα έναν εταίρο ο οποίο αναγνωρίζει πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τι μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό, σημαντικότερο ρόλος που μπορούμε εμεί να διδραματίσουμε να έχουμε τη δέσμευση τη κυβέρνηση. ε, κάτι αρκετά σημαντικό. Ο διάλογο γίνεται ανοιχτά, μπορούμε να του δώσουμε μηνύματα που ε, Συνήθω δια τη διπλωματική οδού θα δίσταζε κανεί να δώσει, αλλά σε μια τέτοια συνεργασία πρέπει κανεί να, να μιλάει ανοιχτά και να ε, συμπεριφέρεται ω πραγματικό φίλο. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε έναν ομολόγο απέναντί μα ο οποίο ακούει, κατανοεί και συνεργάζεται μαζί μα για τη βελτίωση τη κατάσταση. Φυσικά δεν εστιαζόμαστε μόνο στη δημοσιονομική στήριξη. Εργαζόμαστε και σε πιο βασικό επίπεδο με την κοινωνία των πολιτών, ώστε το μήνυμα να διαποτίζει όλα τα επίπεδα, το οποίο ποτέ δεν είναι εύκολο. Και ο επικοδομητικός διάλογος πολιτικής σε χώρες όπως η Ονδούρα, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, ε, επίσης ε, είναι κάτι που εμείς ε, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και ειδικότερα σε τομείς ευαίσθητους όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γενικά θεωρούμε ότι η έκθεση φαίνεται θετική. Να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, αν με επιτρέπετε εδώ η Ονδούρα. Είναι ένας εταίρος όπου όχι μόνο είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τους Ευρωπαίους προλογμένους ε, και όπου η κυβέρνηση εργάζεται, ε, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για αλλαγή, είναι όμως και μια χώρα που δείχνει αλληλεγγύη με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα διεθνή φόρα πριν από μερικά χρόνια σε διάφορα ε, διεθνή φόρα είχαν υιοθετηθεί διάφορες θέσεις και εμείς προωθήσαμε μια θέση υπέρ των κυρώσεων για τις ε, πράξεις της Ρωσίας στην Ουκρανία και η Ονδούρα ήταν μια από εκείνες τις χώρες που ψήφισε μαζί ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που αποτελεί μια αναγνώριση αλληλεγγύης από πλευρά της Ονδούρας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν πιστεύω ότι είναι θετική εικόνα που δίνει η έκθεση Ευχαριστούμε το Ελεκτικό Συνέδριο που λαμβάνει υπόψη αυτέ τι μικρέ χώρε Λατινική Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο, ειδικά ε, με το σημερινό πολιτικό κλίμα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε θέση πλεονεκτική και το γεγονό ότι ε, υπάρχει ενδιαφέρον για μια τέτοια μικρή χώρα, αλλά σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό. Και δείχνει πόσο έθρευστη είναι η κατάσταση σε όλου μα και πόσο σημαντική είναι η μακροχρόνια δέσμευσή μας για τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ όλους σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ντελαρίτση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, συμφωνεί με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ προκειμένου να τις μεταφράσουμε σε επιχειρησιακές δράσεις και πρακτικές. Το σημαντικό για μας είναι ότι η έκθεση αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι καλύτερη μπορεί προκειμένου η Ονδούρα να βελτιώσει το επίπεδο ανάπτυξής της. Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που για μας ε, είναι θετικό. Η έκθεση ε, καταδεικνύει ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εν μέρη αποτελεσματική. Συνεισέφερε σε κάποιες θετικές εξελίξεις, αλλά οι διάφορες συνθήκες στη χώρα, μεταξύ άλλων, ε, παρακολύουν τις ε, ε θετικές συνέπειες. Οι ευρωπαϊκές δράσεις όμως ήταν ε, ουσιαστικές και σε γενικές γραμμές ε, είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις ε, λόγω εξωγενών παραγόντων, αλλά τα αποτελέσματα υπάρχουν. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό για μας ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει στρατηγικές διαλόγου ε, προκειμένου να διαρθρώσει τον πολιτικό διάλογο σε διάφορα επίπεδα στην Ονδούρα και ε, κυρίως σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα που μόλις ε, περιέγραψε και η συνάδελφος. Δεν θα επιμένω σε περισσότερα πράγματα, δύο πράγματα μόνο. Η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να παραπέμψουμε και στην έκθεση η οποία λέει ότι ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντικός και υπήρξε υποχρέωση να δημιουργηθεί πλατφόρμα με την κοινωνία των πολιτών και να υπάρξει νομοθεσία για να βοηθήσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε πώς η βοήθεια και η συνδρομή μας συνέβαλε στις προσπάθειες της κυβέρνησης ε, να αντιμετωπίσει την κατάσταση ε, και ε, η ίδια η Ονδούρα ε, αναγνωρίζει ότι δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση. Κάτι ακόμα θα ήθελα να προτρέψω όλους τους βουλευτές να διαβάσουν το έγγραφο. Είναι μακροσκελές αλλά αξίζει τον κόπο διότι περιλαμβάνονται κάποια πράγματα ε, και εδώ θα είμαι ξεκάθαρος υπάρχουν πάθη στην Ονδούρα μετά από τη δολοφονία ενός ακτιβιστή που ήταν πάρα πολύ σημαντικός και η δολοφονία έγινε πέρσι και υπάρχουν σχόλια παρατηρητών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ε, που ζητούν την αναστολή της βοήθειας ε, επειδή ε, ε, επικρατούν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω ότι η έκθεση αποδεικνύει ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη, διότι τιμωρούμε ανθρώπους οι οποίοι εποφελούνται από αυτή τη συνεργασία. Και πιστεύω λοιπόν ότι αποτελεί καλό ανάγνωσμα αυτή η έκθεση, όχι μόνο για τους βουλευτές, αλλά και για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν τα μέλη μας. Το λόγο έχει ζητήσει πρώτος ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη της Κωνσταντίνα, θα ήθελα να σας πω ότι απαντήσατε πολύ διπλωματικά. Ε, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσάς. Σας ευχαριστώ. Ε, για τον πρέσβη της Ονδούρας γνωρίζετε ότι ε, μια εφημερίδα την περασμένη Δευτέρα, τέσσερις μέρες λοιπόν μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Τραμπ, αναφέρθηκε στις πρώτες απελάσεις ε, στην Ονδούρα. Υπήρξε λοιπόν ένα πρώτο κύμα απελάσεων ε, ελάχιστες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Αυτές είναι οι πρώτες ε, απελάσεις της πολιτικής μετανάστευσης των Πολιτειών. Και ο πρέσβης της Κωνσταρίκας είπε ότι είχαμε κάποια πρώτα σημάδια ότι τα πράγματα ε, θα πάνε καλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προετοιμαζόμαστε των προτέρων. Δεν θα περιμένει ο κύριος Τραμπ να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και άλλωστε ο πρόεδρος, ο κύριος Ερνάντεθ, είπε ότι ε, πρέπει να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τις ευκαιρίες μας αμέσως. Ε, είτε έχουμε νέα εποχή Τραμπ, είτε δεν έχουμε. Δεδομένης λοιπόν και της προστατευτικής πολιτικής που έχει ε, προανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ε, όπως ε, είδαμε στις πρόσφατες δηλώσεις τους, που σημαίνει ότι οι οικονομίες της Κεντρικής Αμερικής που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το επιβεβαιώνουν και διάφορες έρευνες, θα ήθελα να ξέρω τι προβλέπετε για την οικονομία της Ονδούρας. Όπως σας είπα, η οικονομία της Ονδούρας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Αμερικανική οικονομία. Τι προσδοκίες έχετε λοιπόν εσείς μετά από την ανάληψη των καθηκόντων ε, του Τραμπ ε, λόγω και του προστατευτισμού ε, τον οποίο πρεσβεύει. Και επίσης η νέα πολιτική μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι βέβαια νέα κάποια πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες ε, άτομα από την Ονδούρα που έχουν απελαθεί, αλλά δεν θεωρείται ότι θα ενισχυθεί αυτό το κύμα και θα είναι όλα ένα και περισσότερες οι απελάσεις. Σε θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν μπορώ παρά να μη σχολιάσω. Ε, εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει να υποστηρίξουμε την Ονδούρα και την Κεντρική Αμερική εν γέννη και για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν μπορούμε να, να χρηματοδοτούμε και την αντίθετη πλευρά. Περιμένουμε και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά σας. Ε, δεν είναι και όλα ρόδινα στην Ονδούρα βέβαια. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κρίση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρίση η οποία συνεχίζεται και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ονδούρας δεν θέλησε να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας για να συζητήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η διάθεσή μας να υποστηρίξουμε εμπορικά, οικονομικά την Ονδούρα θα πρέπει να σημαίνει και ότι πρέπει να βασιστούμε και σε μία σαφή ε, βούληση, η οποία θα εκφράζεται και σαφώς από πλευράς ε, Ονδούρας να προωθήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην υπάρχουν ε, περιστατικά με υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παρία. Κυρία Τσίνηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για τις παρεμβάσεις σας, ε, για ε, τα όσα είπατε και για την ειλικρίνεια στις παρεμβάσεις σας. Είχα δύο ερωτήσεις, τις οποίες βέβαια με τα όσα είπατε μου τις απαντήσατε ήδη. Μία από τις ερωτήσεις μου ήταν ακριβώς και ήδη δόθηκε απάντηση για ε, το θέμα του συντονισμού των δωρεών ε, και το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες επικαλύψεις. Δόθηκε ήδη μια απάντηση, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέμβουμε και να παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την πτυχή. Το άλλο θέμα ήταν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κύριε Ντελαρίτσε, εγώ θα διαβάσω με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση στην οποία αναφέρθηκατε, αλλά ε, θεωρώ ότι το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ε, η πτυχή αυτή είναι μία από τις ουσιαστικές πτυχές ε, στην οποία θα πρέπει να επιδείξουμε ως Ευρώπη και την παρουσία μας, ε, να υποστηρίξουμε τη δέσμευση και την προσπάθεια της Ονδούρας για να βελτιώσει την κατάσταση μεν, αλλά να στοχεύουμε κυρίως στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ένας ακόμα τομέας ο οποίος αναφέρθηκε και από τον πρέσβη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ο τομέας της καταπολέμησης της διαφθοράς ε, και της καταπολέμησης του εγκλήματος. Ε, διαφάνεια, διαφάνεια στη διοίκηση, διαφάνεια ε, και ορθή διαχείριση ε, των φορολογικών θεμάτων ε, και αντιμετώπιση των οργανώσεων των εγκληματικών που όχι μόνο δημιουργούν ε, ε, προβλήματα ασφαλείας ε, και βίας αλλά έχουν και στόχο την οικονομία των χωρών αυτών. Σε αυτές τις πτυχές λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε κατά την άποψή μου και θα πρέπει να επαγρυπνούμε σε μια απόπειρα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανάπτυξη μεν αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ πολύ. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ μια ερώτηση, απευθυνόμενη στις <clears throat> δύο κυρίες. Άψαμε πολύ μεγάλη προσοχή και τις δύο τοποθετήσεις και η διαπίστωσή μου είναι ότι διαφωνούν στο θέμα της συνεργασίας με τις αρχές. Ε, θα ήθελα ε, λίγες περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορούν να λάβουν ώστε να επιτευχθεί αυτή η θα, θα λέγαμε πολυπόθητη συνεργασία των αρχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάκομσεν πρώτα. Κυρία Γιάκομσεν. Thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εξετάζουμε εμεί το πνευματικότητα τη ενίσχυση τη Ένωση ε, και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ε, Βεβαίω αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολε οι καταστάσει στη χώρα και η βελτίωση παίρνει χρόνο. Όμως ε, για να επανέλθω σε κάποια από τα ζητήματα που ανέφερε ο Διευθυντής το θέμα των στόχων και των βάσεων της βάσης αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει μία βάση, ένα πλαίσιο και στη συνέχεια να έχουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους για να μπορούμε να δούμε την αποτελεσματικότητα. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Όμως ε, είναι σημαντικό για τις διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν να αντιληφθούν ότι για να πετύχουμε κάτι πρέπει να υπάρχουν και στόχοι και κάποιες βάσεις, κάποια πλαίσια. Αυτό θα βελτίωνε τη συνεργασία και με τη διοίκηση. Είμαι βέβαιη, τουλάχιστον από την πλευρά του Ελληνικού Συνεδρίου, ε, εμεί δεν έχουμε προγραμματίσει ελέγχους στη Λατινική Αμερική εδώ και αρκετό καιρό, αλλά είναι σημαντική αυτή η έκθεση διότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια κάποια ορατότητα για την αποτελεσματικότητα των διαφορών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι βέβαιη πάντως ότι επιστρέφοντας ε, στην έδρα μου ε, θα φροντίσουμε να υπάρξει ένα follow-up σε αυτή τη διαδικασία για να δούμε τη βελτίωση και την εξέλιξη στο μέλλον. Είναι θέμα ποικιλομορφίας πολιτιστικής. Ε, λοιπόν, κανείς δεν διαφωνεί με αυτό που λέει το Ελληνικό Συνέδριο και βεβαίως ε, είναι στόχος μας αυτός ε, ε, Εντό εισαγωγικών εμεί διαθέσαμε 8 εκατομμύρια ε, και αντί να βοηθήσουμε τους φτωχούς ε, να ε, δώσουν φαίστη στα παιδιά τους συνεργαζόμαστε με Ινστιτούτα Στατιστικά ε, περνάμε από τους θεσμούς κάνουμε μια προσπάθεια ε, βελτίωσης. Να μιλήσουμε για τους αριθμούς αν θέλετε. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, ε τις, τους εκπροσώπους, τους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους και την ευαισθησία τους. όταν εργάζεται κανείς σε αυτή τη χώρα εμένα μου αρέσει ο πρόεδρος ε, κάνει καλή δουλειά. Ε. Η χώρα ήταν εξαιρετικά εύθραυστη ε, σε θεσμικό επίπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι ήταν ένα failed state, μια χώρα χρεοκοπημένη ουσιαστικά. δεν το ακούει πια κανείς αυτό για την Ονδούρα. υπήρχαν πολύ αρνητικά σχόλια από τους υπερψηφιστές δικαιωμάτων ε, δίνεται μια εντύπωση ότι κάποιοι προσπαθούν να προστατραπήσουν την κατάσταση. Ε, και αυτό βεβαίω καθιστά πολύ σημαντικό το έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά, και από την άλλη ο ρόλο μα ε, πρέπει να είναι προσεκτικό. Πρέπει να δούμε ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να παρέμβουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρετε, σκοτώνεται κόσμο, σκόβουμε ε, την ενίσχυση, τελείωσε. Δεν είναι τόσο απλό. η κυβέρνηση αναγνωρίζει αυτή την αδυναμία που υπάρχει στους θεσμούς, τους, στους της και έχει ζητήσει να δημιουργηθεί ένα όργανο που λέγεται ΜΑΞΙ για την υποστήριξη επακριβώς της, ε, της αντιμετώπισης της ατιμορρησίας ε, και την, ε, για μεγαλύτερη διαφάνεια. Συμμετέχει η οργάνωση Αμερικανικών χωρών, έχουμε χρηματοδοτήσει και εμείς σημαντικά αυτή την προσπάθεια αυτό είναι μεταξύ των βαλίστων πρακτικών. Ε, στην Γουατεμάλα, στην Ονδούρα ε, ζητήθηκε η δημιουργία αυτού του οργάνου και υποστηρίχθηκε η θεσμοθέτησή του. Βεβαίω, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαφθορά, η διαφάνεια, εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία, αλλά πρέπει να, δούμε από πού ξεκινάμε. Έτσι. Δεν ξέρω τα ακριβώ στοιχεία ε, για την Ονδούρα, αλλά ε, φαντάζομαι ότι είναι ο, όπως την υπάρχει την Λατινική Αμερική. Είναι 44, 44 ο δείκτης σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια ε, και τη διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κάτω από το 50 που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Βεβαίως και είναι ένα πολύ αρνητικό στοιχείο και για τις επενδύσεις και για την παρουσία επιχειρήσεων. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις. Δεν είναι εύκολο. Όλοι όμως αντιλαμβάνονται ότι ο, ο δρόμος θα είναι μακρύς και, ότι, και ανηφορικός ε, και εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα για μας αλλά και για την κυβέρνηση ε, να προχωρήσουμε. Θέλω να επιβεβαιώσω προς την Πρόεδρο ότι εμείς συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε σε συντονισμό και με την κυβέρνηση και με τους δωρητές ε, και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αυτός ο κοινός προγραμματισμός από την κυβέρνηση και όλους τους δωρητές εφόσον συμφωνήσουμε γύρω από ένα έγγραφο για το ποιο κάνει τι στη χώρα και θα το βάλουμε αυτό σε ένα χαρτί. Ε, είναι βεβαίω φιλόδοξο αυτό, ιδιαίτερα όταν έχουμε απέναντί μα την Παγκόσμια Τράπεζα ή άλλου τέτοιου εταίρου. Κύριε Πρέσβη, έχετε τέσσερα ολόκληρα λεπτά δικά σα για να κλείσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ θα κάνω σχόλια στις παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει διάθεση για διάφανη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των υπολείπων που συνεργάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τα σχόλιά σας που ακούστηκαν, για τα θέματα αυτά και από την Προεδρία, αλλά διαπίστωσα και κατά την ε, ε, παρέμβασή μου και από την ερώτηση που έγινε στην αρχή. Ε, δεν έγινε συζήτηση με το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα διεθνή θέματα. Δεν ξέρω γιατί δεν συζήτησαν. Ε, είναι αυτή που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία στο χώρα. Ίσως λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος να φανεί ότι υπάρχει και απόλυτο άνοιγμα, αλλά μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Σίγουρα υπάρχει ένα εμπόδιο, ελπίζω όμως να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και ελπίζουμε την επόμενη φορά να υπάρχει παρέμβαση και του Εθνικού Αρμόδιου Φορέα σε θέματα διεθνούς συνεργασίας. Όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριο Φαρία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσετε μια εξαιρετική ευκαιρία. Έχω μια σύνοψη των δύο τελευταίων ετών. Δεν θα σα πω ε, λεπτομέρειε. Ε, ε, θα σα το δώσω στη συνέχεια βέβαια, γιατί πρέπει να είμαι σύντομο. Ε, στις Ονδούρες συστάθηκαν δύο γραφεία για την προστασία ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είπε η κυρία Κινίτσι, και τη διαφάνεια. Υπάρχει το ε, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η αποστολή υποστήριξης της διαφοράς και της ατιμορρησίας. Ε, και οι δύο αυτοί οι οργανισμοί έχουν σαφείς εντολή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπάρχει και μία αναλυτική έκθεση των δύο ετών ε, και των δεσμεύσεων που ανέλαβε και η κυβέρνηση και ο λαός της Ονδούρας ε, για το θέμα αυτό. Υπάρχουν αρκετέ ε, ειδικέ επισκέψεις, τέσσερις από, τα Ηνωμένα Έθνη, δύο από την Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, δύο από τη Διεθνή Διαφάνεια, με έξι πρόοδου ε, που διαπιστώθηκαν και με άλλους οργανισμούς υπήρχαν διάφορες περιοδικές εκθέσεις. Το 2014 είχαμε τέσσερις, το 2015 είχαμε τέσσερις, 2016 τέσσερις, 2017 μέχρι τώρα έχουν γίνει δύο. επομένω αυτά σας δείχνουν με κάποια αριθμητικά στοιχεία λίγο την ουσία ότι ε, υπάρχει πραγματική δέσμευση για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε απλώς τα απαραίτητα και σας λέω ότι εδώ τίθεται θέμα επιβίωσης. Ε, δεν είναι βέβαια απόλυτο, δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω, να πιστοδρομήσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και αυτό ε, καταδεικνύει ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, τώρα ε, δεν ξέρω κάτι για απόρριψη από πλευράς ε, της Προέδρου, του Προέδρου. μπορεί να ήταν στο διεθνές πρόγραμμα του προηγούμενου Προέδρου ή στη γενικότερη ατζέντα που έχουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μην συνομιλήσω με κανέναν και να μην αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά για την επιβεβαίωση, επιβίωση συγγνώμη, της Ονδούρας. Και ε, τέλος, έχουμε και την ερώτηση για το ποιες είναι οι προσδοκία μας ε, με την ε, κυβέρνηση Τραμπ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με το όσα είπε και ο συνάδελφος από την Κώστα Ρίκα. Έχουμε κάποιες θετικές ενδείξεις. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι απελάσεις, ε, κύριε Φαρία, δεν ε, έγιναν από τον κύριο Τραμπ. Υπάρχει μια μακρά απορία πάρα πολλών απελάσεων ε, και από τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση Ομπάμα. Ε, τα αριθμίζουμε σχετικά καλά τα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία ένταξης αυτών των ανθρώπων που επιστρέφουν ε, στη χώρα, στο εργατικό δυναμικό και στον κοινωνικό ιστό. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς έχουμε διαφορετικές συμφωνίες και διαφορετικά καθεστώτα ως ε, κάτοικοι της Ονδούρας και υπάρχουν συγκεκριμένε ε, συνθήκες που καθορίζουν την διαμονή των κατοίκων της Ονδούρας στην ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όχι μόνο τους ε, μετανάστες για λόγους εργασίας, αλλά και σπουδαστές. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ε, συμφωνίες. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο να θεωρήσουμε ότι αυτές οι τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές και από την κυβέρνηση και έχουν εγκριθεί και από το Αμερικανικό Κογκρέσο και την Γερουσία. Και κυρίως ε, υπάρχει και το σχέδιο της Συμμαχίας για την Ευημερία, που υποτίθεται ότι είναι μία απάντηση στη μετανάστευση, δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας, ευκαιρίες υγείας και εκπαίδευσης στις χώρες που βρίσκονται ε, στην Κεντρική Αμερική, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Ελσαβαδόρ. Ε, και υπάρχει υποστήριξη και από το Αμερικανικό Κογκρέσο, ε, και ε, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρξει και κάποια αναθεώρηση αυτών των συμφωνιών. Σαφώς ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθερή δυνατότητα, αν μπορώ να το πω έτσι, και θα δούμε από εκεί και πέρα ε, τι θα γίνει αν υπάρξει μια μαζική μετανάστευση που ελπίζουμε να μην υπάρξει στην Ονδούρα. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η οικονομική μας ανάπτυξη θα πρέπει να φτάσει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να φτάσουμε ε, να έχουμε ευημερία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας πρέπει να υπάρξει και ε, πλήρης συνειδητοποίηση από όλους τους τομείς. Και όταν λέω αυτό τι εννοώ, αναφέρομαι όχι μόνο ε, στο εργατικό δυναμικό αλλά πρέπει να υπάρχει και σε διεθνές πλαίσιο. Ελπίζω να κατάφερα να σας απαντήσω ε, και θα δώσω και αυτές τις εκθέσεις που περιλαμβάνουν και κάποιες προόδους για την διερεύνηση των πρόσφατων εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο θέμα που θα, που θα θέλατε να θέσετε. Δεν υπάρχει. Οπότε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα γίνει στις 27 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Να ευχαριστήσω όσοι παραβρέθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση, τους καλεσμένους μας για τις πληροφορίες που μας παρήχαν και να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε και τους μεταφραστές για την υποστήριξη και για την ανοχή τους όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.